Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε την πράσινη βίβλο για το προσωπικό υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη και να δώσω απευθείας το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής, την Επίτροπο κυρία Βασιλείου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα